Ladies Κυρίες και κύριοι, με λίγη καθυστέρηση, μετά το μεσημεριανό ξεκινάμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Με χαρά υποδέχομαι εδώ την κυρία Ζωελζενή, διευθύντρια εντό τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράση, αρμόδια για πολιτική ασφαλεία και πρόληψη ένοπλων συγκρούσεων. Το θέμα μας σήμερα το απόγευμα είναι οι ζητήματα που σχετίζονται με τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα οι χερσές ε, ε, νάρκες και το έργο iTrace. Ας μην χάνουμε άλλο χρόνο, έχουμε κάποιου χρονικού περιορισμούς, όποτε δυνάμε σωστό λόγο στην κυρία Ζελζενή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ για να σας παρουσιάσω το έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικά σε αυτόν τον τομέα. Θα σας περιγράψω λίγο τα προβλήματα που σχετίζονται με τα όπλα μικρομεγέθους και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα όπλα μικρομεγέθους και τα ελαφρά όπλα. Θα σας αναφέρω κάποια έργα που χρηματοδοτούνται χρυσό αποφάσεων συμπεριλαμβανομένου και του iTrace που αναφέρθηκε στον τίτλο τη συνεδρία αυτή θα σα μιλήσω και για τη συνθήκη Trace ε, μια από τι πιο συναρπαστικέ ε, νομικέ εξελίξει στον τομέα, πιστεύω. Αν σα ενδιαφέρει, θα σα πω και δύο λόγια για το ζήτημα των αυτόνομων όπλων. Θα σας μιλήσω για τις ε, νάρκες και τις σχετικές δράσεις και θα σας πω αν σας ενδιαφέρει και δύο πράγματα για τα χημικά όπλα και τα χημικά όπλα στη Συρία παρότι δεν εντάσσονται αυτά στα φορήτα και ελαφρά όπλα. Ε, αυτά σχεδιάζω να σας πω, οπότε ελπίζω να μείνετε ικανοποιημένοι. Θα έχετε δει τον ειδικό απεσταλμένο για την διάθεση, το Γιάννακ ε, Ζιλιμπεκ. Είχε προετοιμάσει τη διάσκεψη Αναθεώρηση της συνθήκης για τα φορητά όπλα και τον ελαφρύ οπλισμό. Δεν θα σας πω περισσότερα γιατί ο κ. Μπεκά θα επανέλθει στην Επιτροπή εδώ αφού ολοκληρωθεί η διάσκεψη για να σας προσφέρει τα αποτελέσματα της διάσκεψης. Όλοι συμφωνούν ότι από ολόκληρο τον κόσμο μαθαίνουμε τι σημαντικές προκλήσεις ασφαλείας έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εμείς και οι εταίρες χώρε. Ανάμεσα στις διάφορε κακές ειδήσει, τις βιοπραγίες ε, που ακούμε και βλέπουμε καθημερινά είναι τα παράνομα φορητά όπλα και ελαφρύς οπλισμός. Δηλαδή όπλα που παράνομα έχουν περάσει σε τρίτα χέρια, όχι στους αρχικούς αποδέκτες. και που οδηγούν σε πολλούς θανάτους. Είναι ανθρώπινο το ζήτημα, είναι ανθρώπινη απόφαση, η χρήση φορητών όπλων, αυτή είναι η πηγή του προβλήματος, αλλά πολλά μπορούν να γίνουν μέσω δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά σε στενή συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους μας, ώστε να ενισχύσουμε τη διεθνή νομοθεσία, ώστε το εμπόριο των φορητών όπλων να διασφαλίζεται ότι γίνεται νόμιμα και όχι παράνομα. Επίσης, συνεργασία με χώρες εταίρους για να ενισχύσουμε τις δυνατότητες τους ε, αποθήκευσης με ασφαλή τρόπο των όπλων και ελέγχου των ροών όπλων. Πολύ συνοπτικά, αυτό είναι το έργο μας. Αυτά προσπαθούμε να κάνουμε. Εν συντομία να αναφέρω ότι πολλά από τα όσα θα σας περιγράψω χρηματοδοτούνται υπό το CFSP το, για το σχετικό προπολογισμό. Μιλάμε για 17 με 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Για να καταλάβετε αυτό αντιστοιχεί στο 5% του προϋπολογισμού του ε, CFSB. Συνεπώς ε, η μεγάλη πλειοψηφία πηγαίνει σε ε, επιχειρήσεις της κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας και το 5% πηγαίνει την ε, CFSP. Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας. Να σας περιγράψω τα διάφορα έργα τώρα. Σε θέμα νομικής βάσης, νομικής αρχιτεκτονικής, ε, το έργο μας βασίζεται στο πρόγραμμα δράσης των ΗΕ που υιοθετήθηκε πριν από 14 χρόνια και σε, στο Διεθνές Μέσο Ιχνηλάτησης που λατεί τα όπλα και φυσικά έχουμε και την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για Φορητά Όπλα και Οπλισμό του 2005. Θα επανέλθω σε αυτήν. Καλό είναι να ξεκινήσουμε με, μια, με καλά νέα. Την τελευταία δεκαετία, 15 χρόνια, εκατομμύρια όπλα έχουν ανακτηθεί και καταστραφεί. Έχουν δημιουργηθεί καλύτερες συνθήκες ασφαλείας για τις αποθήκες όπλων και πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει νομικά πλαίσια που τους δίνουν τις δυνατότητες για την εφαρμογή καλύτερων πρακτικών στη διαχείριση των όπλων. Οπότε έχουμε ιστορίες επιτυχίας, τις οποίες δεν πρέπει να υποτιμούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει, πιστεύω, σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, να ξεκινήσω με το έργο το δικό μας στις διάφορες χώρες. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα όχι όλα, απλά για να, αποκτήσετε μια, να πάρετε μια γεύση από τη δράση υποστήριξη για τα φορτά όπλα και τον ελαφρύ οπλισμό για παράδειγμα στην Ανατολική Ευρώπη, όπου έχει δοθεί ιδιαίτερη στήση ε, ε, να υπάρξει συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συγκεκριμένες χώρες ε, για να υπάρξει ένας μηχανισμός ελέγχου των φορετών όπλων και του ελαφρύ οπλισμού. Ε, κάποια δουλειά γίνεται σε συνεργασία με τον ΑΣΕ και, την εντύπωση στην ε, Λευκορωσία που πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθεί εστιασμένη στην εκπαίδευση των ελέγχων των εμπορικών ροών και των αποθεμάτων. Ουσιαστικά, αν δεν έχουν αποθηκευτεί ασφαλώς τα όπλα, υπάρχουν δυνατότητες ε, παρεκτροπής τους. Έχουμε δραστηριότητες στη Βόρεια Αφρική και στην ευρύτερη περιοχή του Σαχέλ. Τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου είχαμε υπό τον προϋπολογισμό της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, συνεργασία με τις λιβικές αρχές για τη διαχείριση των ε, αποθεματών όπλων. Δεν θα σα εκπλήξει να μαθαίω ότι έχει ανασταλεί το έργο αυτό δεδομένο των συνθηκών ασφαλεία επιτόπου, αλλά μπορεί να συνεχίσει μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να χάσουμε αυτή την επιλογή την οποία θεωρούμε υψηλή προτεραιότητα. Σε μια χώρα που μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Έχουμε μια άλλη απόφαση του Συμβουλίου στοχευμένη σε διάφορες χώρες του Σαχέλ όπου γίνεται κλασικά ε, η δουλειά που περιέγραψα, συνεργασία με τις αρχές για ενίσχυση του νομοθετικού του πλαισίου και της διαχείρισης των ε, αποθεμάτων όπλων. Έχουμε και άλλη μια απόφαση που αφορά το iTrace ε, και θα επανέλθω σε αυτήν σε λίγο. Έχουμε και άλλα έργα με την ΕΚΟΑΣ, με τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν θα παραθέσω όλα τα έργα αυτά, αλλά ουσιαστικά ε, το σκεπτικό είναι ότι συνεργαζόμαστε με χώρε εταίρου, ενισχύουμε τη δυνατότητά του για τον έλεγχο των μεταβάσεων όπλων, των κινήσεων των όπλων. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για τη δική μα και τη δική του ασφάλεια. Πρόκειται για ένα τομέα όπου η τεχνολογία βρίσκεται υπό διαρκή εξέλιξη, οπότε τα μέσα που χρησιμοποιούμε πρέπει να ακολουθούν αυτή την εξέλιξη. Συχνά από τις χώρες εταίρους ε, ακούμε το εξή σχόλιο, ότι υπάρχει έλλειψη δεδομένων και στοιχείων για το προ τα πού παρεκτρέπονται τα όπλα, πού παρεκτρέπονται τα όπλα από την νόμιμη στην παρανομική κυκλοφορία. Αν δεν έχει κανείς τέτοια στοιχεία, είναι εξαιρετικά δύσκολο να σχεδιάσει αποκρίσεις πολιτικής που να είναι αποτελεσματικές. Ένα από τα πιο καινοτόμα, θα έλεγα, έργα που χρηματοδοτούμε αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας είναι το γνωστό αυτό, το iTrace. Είναι ιδιαίτερα καινοτόμο. Ουσιαστικά χρηματοδοτούμε ανθρώπους που βρίσκονται επί τόπου και διεξάγουν έρευνες και μας αναφέρουν τα όπλα τα οποία έχουν βρει και κατά σχέση, δηλαδή όταν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία και μετά μελετούν αυτά τα όπλα μέσω χνηλάτησης για να δουν σε ποιο σημείο παρεκτράψαν από το νομό εμπόριο. Δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Σαχέλ, στη Συρία και στη Μέση Ανατολή. Ε, τέτοιοι άνθρωποι έχουν καταφέρει να μας προσφέρουν το μεγαλύτερο και πλέον ολοκληρωμένο σύνολο στοιχείων ε, για όπλα στα χέρια του Ισλαμικού κράτους και φυσικά όταν λέω όπλα αναφέρομαι σε όπλα αλλά και πυρομαχικά και σχετικό υλικό λειτουργούν ομαδικά ε, έχουν σωματωθεί στις δυνάμεις Πεσμεργά ε, και βρίσκονται και στη Συρία ώστε να μπορέσουν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει επί τόπου. Τα στοιχεία που αρχίζουν ε, να προκύπτουν ε, δείχνουν ότι η ποσότητα όπλων που έχουν κατασκευαστεί και που έχουν κατασκευαστεί στη ΣΥΠΑ είναι αρκετά υψηλή. Ε, συγγνώμη, είναι αρκετά χαμηλή. Ενώ δεν το περιμέναμε αυτό βάσει των στοιχείων που είχαμε, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα όπλα προέρχονται ουσιαστικά από, στο μεγαλύτερο βαθμό από άλλε χώρε. Αυτή είναι σημαντική πληροφορία. Γιατί όταν θέλει κανεί να δημιουργήσει ένα σύστημα διαχείριση ε, ε, των φορτών όπλων και του ελαφριοπλισμού για να μπορέσει να ελέγξει την παράνομη κυκλοφορία, χρειάζεται αυτή την πληροφορία. Επίση, έχουμε τη συνθήκη εμπορίου όπλων, για την οποία θα μιλήσω σε λίγο την οποία χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε τις αρχές ελέγχου εξαγωγών όπλων ώστε να ανοιχνεύουν την παρεκτροπή των όπλων και να αξιολογούν τους κινδύνους παρακτροπές όταν εξετάζουν άδειες εξαγωγής. Αυτό το στάδιο φυσικά είναι πολύ σημαντικό ε, για να διασφαλίσουμε καλύτερη ε, μεταβίβαση και μεταφορά των όπλων. Θα σα πω δύο λόγια για το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ε, για δράση επί του παράνομου ε, εμπορίου όπλων. Υιοθετήθηκε το 2001 και αποτέλεσε βήμα θεμελιώδης σημασία για να ξεκινήσει αυτή η εργασία μεγαλύτερης εστίασης στην ασφαλή διαχείριση των όπλων. εξακολουθεί να είναι το μόνο διεθνώς νομικά δεσμευτικό μέσο περιλαμβάνει συγκεκριμένες διατάξεις περί υπεύθυνης ε, μεταφοράς όπλων. Μια σημαντική συνάντηση θα γίνει τον Ιούνιο και θα συμμετάσχουμε εμείς πολύ τεχνικής φύσης που θα εξετάσει πολλές από τις πτυχές ε, ε, καλύτερης εχνηλάτησης, εχνηλασιμότητας των όπλων. Επίσης αξίζει να πούμε ότι πολύ σύντομα, στις 13 Μαΐου, θα λάβει χώρα μια συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπό την πρωτοβουλία της Λιθουανίας σε σχέση με το θέμα των ε, φορητών όπλων και του ελαφριού ε, οπλισμού και θα ήθελα να συγχαρώ τη Λιθουανία για αυτή την πρωτοβουλία. Μίλω για τα διάφορα μέσα και τώρα θα μιλήσω σε λίγο για τη συνθήκη εμπορίου όπλων, αλλά ήθελα πρώτα να πω δύο λόγια για τα δικά μας μέσα. Έχουμε τη στρατηγική του 2005 για τα φορητά όπλα και τον ελαφρύ οπλισμό. Θεωρούμε ότι από το 2005 μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλά, οπότε το έγγραφο αυτό ε, χρειάζεται επικαιροποίηση. Ε, να δούμε κατά πόσο χρειαζόμαστε μια επικαιροποιημένη στρατηγική που να, να αντιστοιχεί καλύτερα στις, να καλύτερα στις μεταβολές που έχουν επέλθει στο μεταξύ. Τώρα, η συνθήκη εμπορίου όπλου, όπλων, το λέω και το εννοώ, είναι από τις πιο συναρπαστικές εξελίξεις που είχαμε ποτέ σε θέματα όπλων και όπλων μαζικής καταστροφής, συμβατικών και μαζικής καταστροφής. Είναι εντυπωσιακό ότι επιτευχθεί ε, συνένεση επί του κειμένου. Η συνθήκη εμπορίου όπλων ε, τέθηκε σε ισχύ 24 Δεκεμβρίου πέρυσι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε ρητά τη συνθήκη εμπορίου όπλων και αυτό εκτιμήθηκε ιδιαίτερα. Σήμερα έχουμε 130 υπογράφοντα κράτη μέλη του Ηνωμένων και 67 την έχουν επικυρώσει. Όλα δηλαδή τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων την έχουν υπογράψει και 67 την έχουν επικυρώσει. Είναι μια ιστορία επιτυχίας. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή όσον αφορά την εφαρμογή της συνθήκης εμπορίου όπλων. Φέτος το καλοκαίρι τον Αύγουστο θα λάβει χώρα η πρώτη διάσκεψη, συνάντηση των κρατών ε, που είναι μέρη στη σύμβαση αυτά, όπου θα ληφθούν ορισμένε σημαντικέ αποφάσει, οι οποίε μπορεί να ακούγονται πολύ βαρετέ και τεχνική φύση, γιατί αφορούν ιστορικό κανονισμό, κάποιε διαδικασίε, λήψη αποφάσεων, το που θα βρίσκεται η γραμματεία τη ε, ε, συνθήκη εμπορία όπλων. Τίποτα δεν ακούγεται ιδιαίτερα συναρπαστικό, ωστόσο οι αποφάσεις αυτές ε, θα είναι καθοριστικές για το μέλλον και την αποτελεσματικότητα της συνθήκης ε, εμπορίου όπλων. Αυτή τη στιγμή αυτό παρατηρούμε ότι επειδή δεν υπάρχει συνένεση για το πού θα βρίσκεται η έδρα τη ε, της γραμματείας της συνθήκης εμπορίας όπλων, παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη πολιτικοποίηση των τεχνικών αποφάσεων, αποφάσεων που είναι περισσότερο τεχνικές πρακτικές. Εάν δεν επιτευχθεί κοινή θέση, ο κύριος υποψήφιος, ο πρώτος υποψήφιος είναι Trinidad και τον Πάγκο, με μεγάλη υποστήριξη από πολλές χώρες. Υπάρχουν και άλλοι συναγωνιστές, η Βιέννη και η Γενέβη, όπου υπάρχουν ήδη ε, ε, εγκαταστάσεις ελέγχου όπλων των εθνών. Οπότε αυτό που θα δούμε τώρα μέσα στους επόμενους μήνες θα είναι μια πολιτική συμφωνία, κάποιο είδους συμβασμός ή συνένεση που μπορεί να καταλήξει να είναι εις βάρος της αποτελεσματικής εφαρμογής που αρχικά ήταν ο στόχος μας. Εμείς συνεργαζόμαστε με όλα τα κράτη-μέλη φυσικά ε, Προ υποστήριξη των συζητήσεων για αυτά τα τεχνικά ζητήματα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η συνάντηση του Αυγούστου θα είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Επίσης δραστηριοποιούμαστε ιδιαίτερα στην επαφή με τρίτα μέρη και υποστηρίζουμε τα τρίτα μέρη που θέλουν να δομήσουν το δικό τους νομικό πλαίσιο ώστε να συμμορφωθούν με τη συνθήκη εμπορίου όπλων. Στόχος μας όπως και με τα υπόλοιπα νομικά μέσα παγκοσμίω, είναι ε, το να γίνει, έχει παγκόσμια ισχύ η συνθήκη εμπορίου όπλων. Θέλουμε δηλαδή να ενθαρρύνουμε όσους δεν έχουν υπογράψει να το πράξουν και να συνεργαστούμε με τις χώρες που έχουν υπογράψει ενδιαφέρονται αλλά που ουσιαστικά δεν έχουν τις δυνατότητες να αναπτύξουν ένα εθνικό πλαίσιο τις υποστηρίζουμε. Έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου που εθετήθηκε υπό την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλεία ε, σε συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτό ακριβώ θέλουμε να κάνουμε, να συνεργαστούμε με εταίρου για να αναπτύξουμε τι δυνατότητέ του ε, σύμφωνα με τη, όσον αφορά τη συνθήκη όπλων. Περνάμε τώρα στο θέμα των ε, ναρκών. Οι νάρκε δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δημοφιλέ ως θέμα. Έχει περάσει ο καιρός που ήταν δημοφιλές. Κάποτε είχατε την πρίγκιψα Νταϊάννα που φορούσε ένα κράνος και ένα μπουφάν ε, ασφαλεία και είχε τραβήξει την προσοχή του κοινού, αλλά έχει περάσει πια αυτή η εποχή και σήμερα ο κόσμος ασχολείται με άλλα θέματα που κυριαρχούν στους τίτλους των εφημερίδων αλλά εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το θέμα και θεωρώ ότι δεν πρέπει να το εγκαταλείψουμε διότι είναι μια από τις καλύτερες ιστορίες επιτυχίας που είχαμε ποτέ ξεκινώντας από ένα εθνικό κίνημα ομικρών και διεθνών οργανισμών και καταλήγοντας σε ένα διεθνή μέσο το οποίο σημείωσε τεράστια πρόοδο στον τομέα σε όλο τον κόσμο αλλά δεν πρέπει να χάσουμε την εστίαση. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τις ε, κυβερνήσεις που είναι εταίροι μας να δίνουν προτεραιότητα σε αυτή τη δράση. Και συχνά με ρωτούν γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, δεσμεύει, δεν δεσμεύει ένα ξεχωριστό χρηματοδοτικό μέσο για τη δράση κατά των αρκών. Γιατί την εντάξατε στην κυρία χρηματοδότηση, γιατί δεν υπάρχουν περισσότερες δράσεις, διότι μερικές φορές οι ίδιες οι χώρες εταίροι, παρότι έχουν ακόμα νάρκες, γενικά δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την εξουδετερώση των ναρκών. Αλλά αν δεν προβούμε σε αυτήν, ε, οι επιπτώσεις σε ανθρώπινες ζωές θα αρχίσουν να υπάρχουν. Ε, έχουμε ακροτηριασμούς, ε, νεκρούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν συνεχίζει να είναι, δεσμευμένη. Πήγα πέρσι στο Μαπούτο όπου έγινε η διάσκεψη κορυφή του Μαπούτο, η οποία σήμανε την επέτειο τη συνθήκης τη Οτάβα και όπου είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Υιοθετήθηκε ένα σχεδίο δράσης για τα επόμενα πέντε χρόνια, το οποίο εστιάζεται στην υλοποίηση των δράσεων που έχουν ήδη υιοθετηθεί. πολλές αποφάσεις ε, στη Σύνοδο Κορυφής. Ε, έγινε και μια πολιτική διακήρυξη. Αλλά η ουσία είναι η εξή ότι η διάσκεψη του Μαπούτο και ο λόγος για τον οποίο πολλοί αρχηγοί κρατών και πολλές προσωπικότητες ψηλού επίπεδου πήγαν εκεί είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να ε, μειωθεί η ταχύτητα με την οποία αντιμετωπίζουμε το ζήτημα αυτό. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συμβάλει με πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ μετά από την τελευταία αναθεώρηση της συνθήκης. Ουσιαστικά τι λέμε ότι όταν έχουμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αυτά παρέχουν το 1 τρίτο της ε, χρηματικής ε, ενίσχυσης για αυτό το ζήτημα. Είναι η υπαριθμόν ένα δωρητής. Έχετε, ξέρετε, χώρες σαν το Αφγανιστάν που ήταν από τις χώρες με τις περισσότερες νάρκες στον κόσμο όπου έχουν γίνει το 78% των δράσεων. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τις κυβερνήσει αυτές να δίνουν προτεραιότητα στις δράσεις κατά των ναρκών στα εθνικά αναπτυξιακά τους προγράμματα. Είχα προτείνει να πω δύο λόγια για το ζήτημα των αυτόνομων όπλων και γιατί αποτελεί σημαντικό ζήτημα. Είναι επίμαχο ζήτημα. Δεν υπάρχει κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται υπό εξέλιξη διαρκή. Και ο λόγος για τον οποίο θέλησα να το τονίσω είναι διότι ε, αποτελεί υπενθύμηση ότι η τεχνολογία βρίσκεται υπό διαρκή εξέλιξη και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο μηχανισμός της αντιμετώπισης του αφοπλισμού ε, πρέπει να ακολουθεί τις εξελίξεις. Ε, πρέπει να παρατηρούμε, να παρακολουθούμε πού γίνονται οι συζητήσεις και να βρισκόμαστε εκεί για να διευκολύνουμε τις συζητήσεις μεταξύ των κρατών μελών μας για ορισμένα δύσκολα ζητήματα όπως το τι εννοούμε με τον όρο φωνικά αυτόνομα όπλα γίνεται συζήτηση στη Γενέβη στο πλαίσιο ε, της ε, μιας ενός συστήματος ε, συνθήκης όπλων CCW λέγεται δεν ξέρουμε γιατί ονομαστηκε έτσι πολύ περίπλοκη συζήτηση τι σημαίνει εύλογος αποτελεσματικός ε, ανθρώπινος έλεγχος τι ζητήματα είναι αυτά η προβλεψιμότητα, η αυτονομία και απλά το επισημαίνω ως υπενθύμηση της πολύπλοκης φύσης των ε, θεμάτων με τα οποία ασχολούμαστε Αυτά ήταν τα θέματα που θέλω να σας παρουσιάσω όπως είπα πριν ευχαριστώ να σας πω δύο λόγια για τα χημικά όπλα και για την κατάσταση στη Συρία εάν σας ενδιαφέρει Εκτός ε, μικροφώνου κυρία Πρόεδρος. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη. Όλοι θα γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει στεναρά τη χρήση χημικών όπλων υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Μας ανησυχούν ε, οι επαναλαμβανόμενες καταγγελίες. Είχαμε και πρόσφατα τις καταγγελίες για τη χρήση χλωρίνης ως όπλου ως όπλου στη Συρία. Στέλνουμε ένα πολιτικό μήνυμα αλλά και συγκεκριμένη υποστήριξη της ε, διερευνητικής ε, αποστολής ε, που συστηθήκε για να εξετάσει αυτές τις καταγγελίες, να διερευνήσει αυτές τις καταγγελίες για τη χρήση χημικών όπλων και χλωρίου και εξετάζουμε όλες τις πτυχές ε, για τα χημικά όπλα στη Συρία και στόχος είναι να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι το Συριακό πρόγραμμα έχει τερματιστεί ανεπιστρεπτή. Έχουμε υποστηρίξει ενεργά τον OPCW, ε, τον Οργανισμό για την Απαγόρευση Χημικών Όπλων. Συνολικά 17 εκατομμύρια έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη της καταστροφής των χημικών όπλων που ήταν η πρώτη φάση της επιχείρησης που έχουμε αυτή τη στιγμή. Επιπροσθέτως, αυτή την υποστήριξη δώσαμε για την καταστροφή, πολιτική στήριξη συνεχίζουμε να δίνουμε ώστε να γίνουν οι έρευνες αλλά επιπλέον φυσικά υποστηρίζουμε τον οργανισμό για την απαγόρευση των χημικών όπλων διότι αυτός είναι και ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για τη συνθήκη χημικών όπλων αυτή είναι περιπτώδος άλλη μια ιστορία επιτυχίας είναι το μοναδικό νομικό μέσο το οποίο κατάφερε να διαγράψει μια ολόκληρη κατηγορία όπλων μαζικής καταστροφής η υποστήριξή μας λοιπόν προς τον OPCW αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το 2015 και 2016 θα παράσχουμε 2,5 εκατομμύρια ευρώ προς υποστήριξη των βασικών δραστηριοτήτων του OPCW. Επίσης ένα θέμα που μπορεί να σας ενδιαφέρει γιατί το έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν είναι το ζήτημα της αντιπροσωπείας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των OPCW. Η ΥΠΑΤ εκπρόσωπος ανακοίνωσε την απόφασή της να αναβαθμίσει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των OPCW αποσπώντας έναν αξιωματούχο μόνιμα. Δεν συνέβαινε αυτό στο παρελθόν. Το υποδέχτηκαν θετικά τα κράτη-μέλη και ειδικότερα τα μικρά κράτη-μέλη, τα οποία ξέρετε Εδώ και καιρό ζητούσα να υπάρχει ισχυρότερη παρουσία της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης για να τα βοηθά στις εργασίες. Ε, σκοπός είναι να εδρεύει ο εκπρόσωπος αυτός ε, στο Γραφείο Πληροφοριών στη Χάγη όπου φιλοξενούνται ήδη οι αντιπροσωπείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοινοβουλίου. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Και νομίζω ότι εδώ μπορώ να ολοκληρώσω την ομιλία μου. Πολύ ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, παρόλο που είναι εξαιρετικά σημαντικό το θέμα αυτό και ενδιαφέρον, Δεν ε, μπορούμε ακόμα να επικροτούμε και να πανηγυρίζουμε. Πρέπει εμείς να το αξιολογήσουμε. Δεν θα μιλήσω παραπάνω για να έχουν τα μέλη την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις. Θα ήθελα ωστόσο να σας ε, ρωτήσω για τη Βοσνία Ερσεγοβίνη και για την κατάσταση εκεί με τα αποθέματα των όπλων και την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, αυτό που μας ε, ανησυχεί είναι τα περιφερειακά όπλα μικρού διαμετρήματος ή φορητά. Αν δεν υπάρχει λαθρεμπόριο, σίγουρα υπάρχει εμπόριο τέτοιου είδους όπλων σε διάφορες περιοχές οι οποίες πολλαπλασιάζονται. στι παρυφές των ευρωπαϊκών συνόρων. Πώς αξιολογείται ε, το εργαλείο ε, iTrace Βέβαια δεν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μπορείτε να μας κάνετε μια σύντομη αξιολόγηση του iTrace. Ποια είναι τα σχέδιά σας. Πώς θα ενισχύσετε την επιχειρησιακή του δυνότητα. Πιστεύετε ότι μπορούμε να καλύψουμε τις περιοχές μας. Έχουμε αυτή την ικανότητα. Άκουσα την παρουσίασή σας με μεγάλο ενδιαφέρον και είδα ότι Η παρακολούθηση των όπλων μας δείχνει ότι η προέλευση των όπλων δεν είναι η συνηθισμένη, δεν είναι αυτή που θα νόμιζε κανείς. Δεν είναι κατά κύριο λόγο η ΙΠΑ. Ξέρετε, παλιά λέγαμε δεν είναι η Αμερική, αλλά δεν λέγαμε από πού ή ποιες είναι οι άλλες δυνατότητες σε σχέση με τη δική μας περιοχή. Αυτά έχω εγώ να πω, αλλά θα ήθελα να καλέσω και άλλα μέλη να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Πανστροζιεύσκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πριν από πολλά χρόνια αναφέρατε ότι υπήρχε τεράστιο πρόβλημα με διαφόρων ειδών νάρκες. Ξέρω ότι πολλές ε, χώρες έχουν υποσχεθεί να τις καταστρέψουν με διάφορα χρονοδιαγράμματα και με διάφορες προθεσμίες. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, γιατί ξέρω ότι οι νάρκες από την Ευρώπη φτάνουν στην Αφρική. Συγγνώμη, επειδή έπαιζα με τα ακουστικά μου δεν άκουσα την αρχή της ερώτησης. Μπορείτε να μου την ξαναπείτε. Ναι, βεβαίως μπορώ να σας ε, την ξαναπώ. Ή ξέρω ότι όπλα και ειδικότερα νάρκες διοχετεύθηκαν στην Αφρική πριν από κάποια χρόνια. Και τα ευρωπαϊκά κράτη υποσχέθηκαν να τις αφοπλίσουν, να τις καταστρέψουν αυτές τις νάρκες. Που ήταν σε απόθεμα αχρησιμοποιητές για πάρα πολλές δεκαετίες. Έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Έχετε πλήρη έλεγχο της διαδικασίας. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε και άλλους. Και αν δεν υπάρχουν, σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω με τη Βοσνία. Και χαίρομαι που μου θέσατε αυτό το ερώτημα. Είναι μία από τις χώρες στις οποίες πέρασα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του πολέμου και όντως η νάρκες ήταν πολύ σημαντικό πρόβλημα εκεί στη Βοσνία το USCE έχει την πρωτοκαθεδρία στην προσπάθεια εξουδετέρωσης και εφοπλισμού των ναρκών. Υπάρχουν μη, μη σταθερά, ασταθή πυρομαχικά που πρέπει να καταστραφούν και πάρα πολλά αποθέματα που πρέπει να καταστραφούν. Η πρόοδος δεν ήταν όσο, τόσο γρήγορη όσο θα ήλπιζε κανείς ιδανικά και τολμώ να πω ότι δεν είναι αυτός ο μόνος τομέας όπου η πρόοδος δεν ήταν τόσο ταχεία όσο θα ήλπιζε κανείς. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουμε να επενδύουμε σε αυτό το πρόγραμμα που ανέφερα προηγουμένως. Το πρόγραμμα CSAC, Clearing House Program. Το CSAC λοιπόν παραμένει σαν πρόγραμμα και ενεργό και συνεχίζει να εκτελείται στη Βοσνία είναι ένα πεδίο όπου θα, χρειαστούν, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Τώρα ως προς το iTrace. Όντως βρισκόμαστε στις αρχές του. Το είπατε κι εσείς. Δεν είναι ένα έργο που υλοποιείται εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Όμως η αρχική αξιολόγηση είναι πολύ θετική. Θετικό είναι το πρόσημο και στις αντιδράσεις και στις απαντήσεις που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη και από τους εταίρους. Όλοι, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι εξαιρετικά θετικά έναντι αυτού. Ξέρω ότι υπάρχει κάπου το, ακριβώς, το ακριβές νούμερο των υποθέσεων που έχουν διερευνηθεί σε σχέση με όπλα, τα οποία, ε, για τα οποία συνεχίζεται βέβαια η έρευνα. Θα το βρω το νούμερο εντός ολίγου. Εν πάση πτώση, ε, στο επίκεντρο βρίσκεται το εξής. Σας ευχαριστώ Κλάρα είναι η επικεφαλής ε, της ε, διεύθυνσης ε, της οποίας προείσταμε για τη μη διάδοση των όπλων και των αφοπλισμών και υπέρ του αφοπλισμού κτλ. Λοιπόν, 100.000 όπλα έχουν καταγραφεί, 100.000 όπλα πυρομαχικά και σχετικό υλικό σε 8 χώρες που έχουν πληγεί από τις συγκρούσεις είναι πολύ περισσότερα από ό,τι έχει ερευνηθεί από οποιοδήποτε άλλο όργανο, εργαλείο, πρόγραμμα που έχει ως αντικείμενο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου όπλων. Ε, και εντοπίζουν τα στοιχεία από πρώτο χέρι, αλλιώς δεν τα απελευθερώνουν ούτε τα διαδίδουν. Μιλούμε για 100.000 όπλα πυρομαχικά κτλ. Και, και είναι στοιχεία που έχουν βρει οι ίδιοι, δεν τα έχουν δεχθεί από άλλους, ούτε είναι από δεύτερο χέρι. Είναι εξαιρετικά επιφυλακτική και προσεκτική. Είναι οι πιο προσεκτικέ προβλέψει. Παρ' όλα αυτά φτάνουμε στο νούμερο 100.000. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε διαδικτυακή τοποθεσία και έτσι οι εταίροι μπορούν καλύτερα να εντοπίσουν, να αντιληφθούν το πρόβλημα και να πάρουν τα μέτρα, τα απαραίτητα για ε, να αποφευχθεί η παρεκτροπή της χρήσης. Είναι σημαντικό να επεκταθεί το πρόγραμμα iTrace σε μια δεύτερη φάση, σε ένα δεύτερο χρόνο. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλή ιδέα. Τα κράτη-μέλη εκδηλώνουν το ενδιαφέρον να δοθεί παράταση στο πρόγραμμα αυτό, ωστόσο δεν είναι βέβαιο θα είναι αντικείμενο συζήτηση για τους επόμενους μήνες. Τώρα μας ρωτήσατε ποιες χώρες ευθύνονται για την ε, εκτροπή, την ε, ε, παράνομη χρήση αν θέλετε. Δεν έχω όλο τον κατάλογο χωρών μπροστά μου, αλλά από μνήμης μπορώ να σας αναφέρω τις χώρες της Αφρικής, στην αρχή πρώτη στη λίστα το Σουδάν, μετά Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, που τελικά είναι μια χώρα η οποία δεν έχει πληγεί τόσο πολύ από τις συγκρούσεις, ε, ωστόσο υπάρχουν προβλήματα ασφάλειας. Είναι χώρες που εν μέσω εμφυλίου πολέμου είχαν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έπληξαν τις ίδιες, αλλά έπληξαν και τη δική μας ασφάλεια όπως γνωρίζετε. Άλλες χώρες που ε, βρίσκονται ψηλά στη λίστα αυτή είναι η ακτή του ελεφαντοστού, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, η Συρία, το Δυτικό Ιράκ, το Βόρειο Μαλί και το Τσάντ. Βέβαια, έχει χειρή παρουσία. Επίσης, το ερώτημα για τις νάρκες και κατά πόσο προορίζονται και κατευθύνονται στην Αφρική. Δεν ξέρω αν σας κατάλαβα καλά. Μιλήσατε για πρόσφατες μεταφορές ναρκών από την Ευρώπη στην Αφρική. Δεν, πολύ ότι δεν το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από τις δικές μας πληροφορίες και από τα δικά μας στοιχεία, τα περισσότερα από θέματα ναρκών στην Αφρική πράγματι έχουν καταστρα... καταστραφεί. Είναι μια ιστορία προόδου. Δεν θα πω success story, δεν θα πω ιστορία επιτυχίας, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, progress story ιστορία προόδου, γιατί έχει σημειωθεί προόδος σημαντική στην καταστροφή των αποθεμάτων ε, ναρκών. Ωστόσο, ορισμένα ναρκοπαίδια δεν έχουν ακόμα εξουδετερωθεί σε αρκετές χώρες, π.χ. στην Αγγόλα, μια άλλη χώρα στην οποία ε, έχω ζήσει και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι συνεχίζουν να υπάρχουν ναρκοπαίδια εκεί. Το ίδιο και στη Ζιμπάμπουε. Κάποιες άλλες χώρες επίσης περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατάλογο και έχουν τεράστιες ανάγκες. Και πρέπει να συζητήσουμε σε ποιο βαθμό ε, θα είμαστε σε θέση να στηρίζουμε αυτό, αυτή την προσπάθεια εξουδετέρωσης των αρκών στα υφιστάμενα ναρκοπαίδια. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Θα έλεγα ότι μπορεί ίσως να υπήρξε από πλευράς διερμηνίας ε, ένα ζήτημα σε σχέση με την τοποθέτησή σας. Νομίζω ότι υπήρξε κάποια παρανόηση με άλλα λόγια στην αρχή αρχή της ερώτησης. Μήπως θα θέλατε να επαναλάβετε την ερώτηση, να εξειδικεύσετε. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την ευκαιρία αυτή. Διότι η ερώτησή μου <clears throat> βασιζόταν στην προηγούμενη εμπειρία μου στο Πολωνικό Κοινοβούλιο ήμουν επικεφαλής μιας επιτροπής αρμόδιας για την εθνική άμυνα. Κάπου μια δεκαετία πριν οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν υποσχεθεί να καταστρέψουν αυτές ε, τις νάρκες ώστε να σταματήσει το παράνομο εμπόριο και η διακίνηση, παράνομη διακίνηση ναρκών προς την Αφρική ουσιαστικά και μη ευρωπαϊκές χώρες προσυπέγραψαν αυτή τη συμφωνία. Είναι σημαντικό να στεφθεί με επιτυχία αυτό το εγχείρημα ο όγκος των ναρκών που διοχετεύεται προς την Αφρική, ο αριθμός πάγωσε ή μείωσε συνολικά. Η ερώτησή μου όμως ήταν διαφορετική. Ο έλεγχος καταστροφής των ναρκών παγκόσμια όσον αφορά τις χώρες προέλευσης αυτών των όπλων. Ολοκληρώθηκε αυτό το εγχείρημα. Βρισκόμαστε πραγματικά, έχουμε έλεγχο της καταστροφής των ναρκών και τι συμβαίνει. Μάλιστα. Και μία πτυχή που κατά τη διάρκεια της δικής μου θητείας στο Πολωνικό Κοινοβούλιο συμμετείχα στην ε, ε, επικύρωση της σύμβασης ε, από την Πολωνία και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η χρήση ακριβώς ως πτυχίο, ήταν ένα πολύ σημαντικό θέμα που βρέθηκε υπό συζήτηση Θεωρώ λοιπόν ότι η κύρια πτυχή αυτού του ερωτήματος ήταν ακριβώς αυτή η πτυχή της χρήσης, η παράμετρος της χρήσης. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Όπως προανέφερα, όσον αφορά την καταστροφή αποθηκευμένων όπλων, έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος και σχεδόν όλες, όλα τα αποθηκευμένα αυτά όπλα στην Αφρική σχεδόν έχουν καταστραφεί. Υπό τον, τους όρους του εμπορίου ναρκών είναι κάτι που έχει σταματήσει. Περί αυτού επρόκειτο με τη συνθήκη της ε, Όταβα του Καναδά. Δεν γνωρίζουμε εμείς ε, με κανένα τρόπο για κάποιο εμπόριο ναρκών που να βρίσκεται υπό εξέλιξη. Δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες, δεν έχουμε γνώση για κάτι τέτοιο. Και αυτό πάλι αποτελεί τμήμα της επιτυχίας, της επιτυχίας με την οποία στέφθηκε η σύμβαση της Οτάβας του Καναδά. Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία. Τώρα, παιδεία ναρκών ή ε, εκεί όπου απομένουν και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι καταστροφές ε, ναρκών ε, που πρόκειται να μπορέσουν να εξουδετερωθούν σε σχέση με την περίοδο που είχαν στη διάθεσή τους οι χώρες για την καταστροφή των ναρκών. Υπάρχει το αίτημα το οποίο έχει διατυπωθεί για την παροχή συνδρομής βοήθειας για να συνεχιστεί η αποναρκοθέτηση και η καταστροφή των ναρκών και ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα αυτά. Κυρία, θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα, το θέμα της Ουκρανίας οι διατάξεις της συμφωνίας του Μίνσκ είναι η Ουκρανία να έχει τον έλεγχο, απόλυτο έλεγχο των συνόρων της χώρας συνολικά. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι οι παραβιάσεις της συμφωνίας του Μίνσκ συνεχίζονται, βρίσκονται υπό εξέλιξη και σημειώνονται παραβιάσεις και παραβάσεις και μεγάλες συγκρούσεις διεξάγονται γύρω από τη Μαριούπολη για παράδειγμα, πράγμα το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Και όπως γνωρίζουμε η Ουκρανική κυβέρνηση μας λέει ότι η Ουκρανία είναι ας το πω έτσι πεδίο βολής ή πεδίο δοκιμών σύγχρονο, σύγχρονου ε, και μάλιστα πολύ ε, ε, ε, προηγμένου οπλισμού από πλευρά των Ρώσων, ποιες δυνατότητες έχετε να ελέγχονται αυτέ οι ροέ όπλων εκεί τώρα, αυτή τη στιγμή. Ποιες είναι οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της δική σας υπηρεσίας, πώς να το πω, της δικής σας μονάδας ή της, του δικού σας τμήματο για να εποπτευθεί αυτή η υπόθεση. Να παρακολουθήσετε δηλαδή την κατάσταση εκεί εκ του σύνεγγης και ποιες δυνατότητες υπάρχουν με άλλα λόγια για να μπορέσει κανείς να έχει μια αξιόπιστη παρακολούθηση και εποπτεία των όσων τεκταίνονται εκεί. Γνωρίζω ότι δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα οι επόπτες ε, ε, παρατηρητές του όσα αλλά θα πρέπει να δοθεί υποστήριξη ώστε να συνεχιστεί η εποπτεία. Θα θέλαμε να σταματήσουν δηλαδή οι ροές όπλων προς αυτή την περιοχή, προς τμήματα της επικράτειας της Ουκρανίας. Θα θέλατε να σχολιάσετε επ' αυτού, παρακαλώ. Αναερώτηση θα προσπαθήσω να απαντήσω και θα ε, ζητήσω πρώτα από την κυρία να τοποθετηθεί, μετά θα λάβετε εσείς τον λόγο. Για την Ουκρανία λοιπόν που αναφέρατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πράγματι σφόδρα τα μάλα των ΟΣΑ για να υπάρξει αυτή η παρακολούθηση. Αυτός είναι ο κύριος διάβλος και επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα με βάση τις διατάξεις της συμφωνίας ε, της σύμβασης του Μίνσκ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική λύση που θα εξευρεθεί για αυτό το ζήτημα και ιδιαίτερα υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για την αποτελεσματική πλήρη εφαρμογή αυτών των διατάξεων αυτής της συμφωνίας. Υπήρξε συγκεκριμένο αίτημα τώρα της ε, Ουκρανίας αλλά δεν υπάρχει κάποια θέση που να έχει ληφθεί κάποια απόφαση για επιπρόσθετη ε, βοήθεια και σύνδρομη. Ο κύριος ε, Πρόεδρος Τάσκα... Ντόναλτ Τούσκ είπε ότι θα το εξετάσει. Είναι μια δυνατότητα παροχής ε, αυτή η βοήθεια για τα μελήματα αυτά που αναφέρθηκαν. Ευχαριστώ. Η δική μου όμως αναφορά ήταν σε σχέση με κάποια στοιχεία τα οποία υπάρχουν και για τις συζητήσεις ε, που βρίσκονται υπό εξέλιξη στο Κοινοβούλιο. Φυσικά γνωρίζουμε το αίτημα που διατυπώθηκε από την Ουκρανία. Αναζητούνται όμως δυνατότητες για να ενισχυθεί η εποπτεία από πλευρά όσα μετά από την ε, αποστολή ε, στην Ουκρανία θεωρούμε ότι θα πρέπει ίσως να θεωρηθεί αναγκαίο, επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί αυτή η εποπτεία από πλευρά του ΩΣΑ. Θα θέλαμε τη δική σας άποψη. Το θεωρείτε και εσείς αναγκαίο να ενδυναμωθεί αυτή η δραστηριότητα του ΩΣΑ των ε, εποπτών των παρατηρητών με μεγαλύτερους αριθμούς και δυναμικό από πλευρά τους. Απάντηση. Θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει στον ΩΣΑ να προσφερθεί αυτή η υποστήριξη για τους παρατηρητές επόπτες και σίγουρα υπάρχει, ε, για τον ΟΑΣΕ με συγχωρείτε, υπάρχει σίγουρα η βούληση και η χορήγηση, ε, για τη χορήγηση αυτής της ε, συνδρομής θωρακισμένα οχήματα για παράδειγμα που μπορούν να διατεθούν δορυφορική εποπτεία ε, όλα αυτά βρίσκονται υπό εξέλιξη ως μέτρα συνδρομής από πλευράς του ΟΑΣΕ και θα ήθελα να πω ότι υπάρχει εδώ και η δυνατότητα να παράσχουμε τη συνδρομή μας με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουμε να καταστρέψουμε τις ε, νάρκες που ε, βρίσκονται εκεί και, έχουν, και βρίσκονται και σε αποθήκες ώστε να μπορέσουμε είτε από πλευράς ΝΑΤΟ και δικής του δράσης να δούμε. Βρίσκεται υπό εξέλιξη η συζήτηση με τις ε, αρχές της Ουκρανίας, με την ε, Ουκρανική κυβέρνηση για τέτοιου είδους δραστηριότητες και αυτό αποτελεί τμήμα ενός ε, εύρους μέτρων, μιας δέσμης μέτρων που μπορεί να παρασχεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς υποστήριξη της Ουκρανικής κυβέρνησης. Επιπρόσθετα σε ένα μεγάλο εύρος μέσων και εργαλείων που θα μπορούσαν να παρασχεθούν για ένα ολόκληρο, ολοκληρωμένο πλαίσιο αβοήθειας και συνδρομής προς την Ουκρανία. Ο κύριος Σαφχάουζερ, παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι ερώτηση ουσιαστικά. Εγώ έχω πάει ο ίδιος στο Ντονέτσκ προσώπος, και έχω να σας πω ότι οι νάρκες ε, κατά προσωπικού που σκοτώνουν παιδιά χρησιμοποιούνται από το Κιέβο. Το ίδιο και οι νάρκες ε, διασποράς ε, σε αυτές οφείλονται χιλιάδες ε, νεκροί η κυβέρνηση του Κιέβου έχει στραφεί κατά του λαού της Ουκρανίας με επιπλέον όπλα που απαγορεύονται στις συμβασίες της Γενέβης. Εγώ είχα την ευκαιρία να συναντήσω παιδιά που ακροτηριάστηκαν εξαιτίας αυτών των αρκών. Επίσης, θα ήθελα να σας πω για τις συμφωνίες του Μίνσκ. Πρέπει να είμαστε ακριβείς θα πρέπει να τις γνωρίζετε, τουλάχιστον το ελπίζω. Η πλήρης αναγνώριση των συνόρων της Ουκρανίας αποτελεί απόλυτη αρχή, πράγματι. Αλλά η διαδικασία αυτή θα μπορέσει να εφαρμοστεί και αυτό αναφέρεται στις συμφωνίες του Μίνσκ μόνο όταν η κυβέρνηση του Κιέβου θα έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις τοπικές κυβερνήσεις του Ντόνατσκ και του Λουγκάνσκ για να συμφωνήσει επί μιας διαδικασίας αποκέντρωσης αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του Κιέβου δεν έχει ξεκινήσει τέτοια ε, διαπραγματεύσεις. Όλοι οι παρατηρητές ε, του ΟΑΣΕ και οι τοπικοί παρατηρητές ε, συμφωνούν επ' αυτού. Η κυβέρνηση του Κιέβου λοιπόν δεν μπορεί σύμφωνα με τις συμφωνίες του Μίνσκ να αποκτήσει ακέραια σύνορα γιατί δεν έχει ακόμα ξεκινήσει να αναλάβει ευθύνη το συνόρο του επειδή δεν έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσει με τι ε, κυβερνήσει του Ντονέτσκα και του Λουγκάνσκα. Κύριε Σαφχάουζερ, πρόεδρο, αντιλαμβάνομαι ότι το περιεχόμενο τη συμφωνιών του Μίνσκ δεν είναι το θέμα τη σημερινή συνεδρίαση. Αναφερόμαστε τώρα στην παρακολούθηση της ροή ε, των ροών όπλων. Το θέμα είναι η μη διάδοση και ο αφοπλισμός. Σίγουρα αυτά που είπατε για τις νάρκες ε, έχει σχέση με, έχουν σχέση με το ζήτημα, αλλά παρακαλώ εστιαστείστε στο θέμα της συνεδρίας αυτής. Θέλουμε να μιλήσουμε και για το iTrace. Ευχαριστούμε. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Mrs. Would you like Κύριε Ζενή, θέλετε να μιλήσετε για το θέμα αυτό. Ε, σημειώνω τα όσα είπατε. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι δεν έχουμε δει καμία επαληθευμένη έκθεση που να δίνει οποιαδήποτε πληροφορία περί χρήσης ναρκών από την Ουκρανική κυβέρνηση. Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, δεν υπάρχουν πληροφορίες, ε, δεν έχουμε δει καμία έκθεση που να σύμφωνη με τα όσα είπατε. Uh, Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Πιστεύω ότι έχουμε ολοκληρώσει αυτό το κομμάτι της συνεδρίασης. Να ευχαριστήσω την κυρία Ζελζενή για αυτή την πολύ ε, ενημερωτική και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ενημέρωση. Ε, ξέρετε, η συνάντησή μας τώρα λαμβάνει χώρα παράλληλα με σημαντικές ψηφοφορίες ε, στο Κοινοβούλιο, σε άλλες επιτροπές, οπότε δεν είχαμε μεγάλη συμμετοχή και προσέλευση, αλλά σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ακριβώς στις 4 και 30 θα έχουμε το νέο Γενικό Διευθυντή της EDA, τον κύριο Χόρχε Ντομέκ. Οπότε παρατηρώ, παρακαλώ μην φύγετε και θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση στις 4.30. Να ευχαριστήσω την κυρία Ζελζενή και την κυρία Κλάρα Γκάσλεν που ήταν ήδη παρούσα στην πρωινή μας συνεδρίαση. και μας παρουσίασε τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστούμε.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 Ladies Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Χόρχε Ντόμεκ, εκτελεστικό διευθυντή της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Αμήνης. Ο κύριος Χόρχε Ντόμεκ μου είπε ότι σήμερα είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συναντάτε με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι συμμετείχε το πρωί στο πρωινό γεύμα εργασίας που οργάνωσε ο κύριος Γκάλαχερ με αντικείμενο παρεμφερεί ζητήματα, τα ίδια ζητήματα. Αυτό είναι καλό. Επομένως είμαστε έτοιμοι να το ξανασυζητήσουμε. Άλλωστε το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό εν ώψη του, της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου, η οποία θα ασχοληθεί και με τις ευρωπαϊκές αμυντικές ικανότητες, δυνατότητες, τρέχουσα κατάσταση των εξελίξεων. Σίγουρα το ίδιο ζήτημα θα συζητηθεί και σε επίπεδο Υπουργών Αμήνης και θα υπάρξει ενημέρωση και αποτίμηση των πεπραγμένων. Όμως, για πρώτη φορά Ο νέος εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας έρχεται στη δική μας υποεπιτροπή για την ασφάλεια και την άμυνα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση που μου απευθύνατε σήμερα. Χαίρομαι ιδιαίτερος διότι μπορώ να πάρω το λόγο στην Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Αμήνης για πρώτη φορά με την νέα ιδιότητά μου του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας. Από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, έχω μεταβεί στις περισσότερες πρωτεύουσε των κρατών μελών για να προσπαθήσω να καλλιεργήσω ένα, μια αίσθηση ιδιοκτησίας από πλευράς κρατών μελών, να μοιραστώ μαζί τους το, όραμά μου για τους μελλοντικού προσανατολισμούς της υπηρεσίας και θα ήθελα σήμερα να έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με εσά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Εκτιμώ ιδιαίτερα στην αλληλεπίδραση που έχουμε και θέλω να διατηρηθεί και να παραμείνει. Η ομιλία μου θα κινηθεί γύρω από τρει άξονε. Πρώτον, την άποψή μου για το ρόλο τη υπηρεσία στο μέλλον. Δεύτερον, προετοιμασία για τη Σύνοδο Κορυφής ε, του Ιουνίου. Και τρίτον, ενημέρωση για τα προγράμματα τα αμυντικά ε, απόκτησης αμυντικών ικανοτήτων τη Ευρωπαϊκή Αμυντική Υπηρεσία. Α ξεκινήσω με το όραμά μου για την υπηρεσία αυτή για το μέλλον. Καταρχάς, Θεωρώ ότι η υπηρεσία αυτή είναι μια υπηρεσία διευκόλυνσης, είναι ένας παράγοντος που θα διευκολύνει και θα βοηθήσει στην επίτευξη των φιλοδοξιών των κρατών μελών. Είναι βασικός μας ρόλος να στηρίζουμε τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν βασικές ικανότητες και θα πρέπει να είναι διαρθρωμένες, δομημένες αυτές οι ικανότητες οι αμυντικές, να τους επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε περαιτέρω ευρωπαϊκή αμυντική ολοκλήρωση. Η αναθεώρηση ε, του σχεδίου ε, για την ανάπτυξη ικανοτήτων της υπηρεσίας θα είναι και ο βασικός μοχλός να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Από εκεί και πέρα, στόχος μας είναι όχι η οργάνωση ασκήσεων ε, με αυτό σκοπό να έχουμε ασκήσεις. Αυτές οι δραστηριότητες θα πρέπει να συμβάλλουν στο να γίνουν πιο ισχυρές οι ικανότητες αυτές οι αμυντικές Έχουμε το πρόγραμμα για την άσκηση των ελικοπτέρων που επέτρεψε να ωφεληθούν από πολυεθνική κατάρτιση περίπου 12.000 στρατιωτικοί οι οποίοι έχουν ξανασυναντηθεί σε διάφορα σκηνικά επιχειρήσεων ανά τον κόσμο. Η ετήσια άσκηση για την αερομεταφορά μας έκανε να εξοικονομήσουμε περισσότερα από 500 500,000. για 500.000 ευρώ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε και ε, ευρωπαϊκά κονδύλια για την ε, χρηματοδότηση της έρευνας σε θέματα αμυντικά. Συμπληρώνουμε την εθνική έρευνα. Λειτουργούμε συμπληρωματικά. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να, να διατηρήσει την αυτονομία της. Εάν δεν αναλάβουμε ε, δράση, η αμυντική και τεχνολογική βιομηχανική βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα φθήνει και θα, έχουμε, θα διατρέξουμε τον κίνδυνο να γίνουμε μια ήπειρος υπεργολαβιών. Και αυτό θα έχει επίπτωση και στην ανάπτυξη και στην αποσχόληση να μην λησμονούμε ότι οι βασικοί εργολάβη σε δραστηριότητες στρατιωτικές και πολιτικές έχουν παραμείνει σε ευρωπαϊκό έδαφος μέχρι σήμερα διότι ε, προμηθεύουν ε, MODs. Και δηλαδή Υπουργεία Μήνης, Ministries of Defense, MODs. Η προστιθέμενη αξία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας είναι σαφέστατη. Μπορούμε να μετριάσουμε τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών κανονισμών για τα αμυντικά για να μην πληγούν οι αμυντικές ικανότητες των κρατών μελών. Μπορούμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά κονδύλια, διαρθρωτικά ε, ε, ε ταμεία, πρόγραμμα COSME για να ενισχύσουμε την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Υπηρεσία στηρίζει και τα κράτη-μέλη που συμμορφούνται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ε, για τα θέματα τη οδηγία REACH, για παράδειγμα, αλλά και για τα θέματα των δημοσίων αγορών ή κρατικών προμηθειών. Και οι ιδιαιτερότητε ε, των αμυντικών θεμάτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στι ευρύτερε ευρωπαϊκέ ε, πολιτικέ και η EDA, η υπηρεσία μα, το λαμβάνει υπόψη αυτό. Εξαιρετικό παράδειγμα είναι το Single European Sky, ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός. Και έχουμε και το Σέσαρ το Caesar και Σαρά στο πρόγραμμα που είναι το τεχνολογικό σκέλος έτσι ώστε οι στρατιωτικές δυνάμεις να έχουν ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση στα αέριους χώρους για θέματα κατάρτισης, εκπαίδευσης και ούτω καθεξής. Στόχος της υπηρεσία μας είναι να διατηρήσει η ικανότητα, την ικανότητά του, να διατηρήσουν οι εκάστοτε ένοπλες δυνάμεις ευρωπαϊκές την ικανότητά τους να παρεμβαίνουν στο διεθνές στερεώμα, να μπορούν να είναι ε, ε, μάχημες, να μπορούν να αναλάβουν δράση. Και ε, σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε και στη διαχείριση της εναρίας κυκλοφορίας με ασφαλή τρόπο και μάλιστα σε τα, με τακτό χρονικά τρόπο. Έρχομαι τώρα ε, στο δεύτερο άξονα της ομιλίας μας, την προ ομιλίας μου την προετοιμασία για τη Σύνοδο του Ιουνίου. Ελπίζω περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν οι ηγέτες ε, στα θέματα μήνυσης σε σχέση με το 2013. Άλλωστε πολλά πρέπει να συζητηθούν. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν μπορεί ε, να είναι μια άσκηση κατά την οποία απλά γίνεται αποτίμηση των εξελίξεων. Θα πρέπει να δοθεί όθηση από υψηλό πολιτικό επίπεδο προς τα κάτω. Ε, η στρατηγική για την ασφάλεια είναι ένα πολύ πολύτιμο εργαλείο. Ωστόσο η στρατηγική, όσο καλή και αν είναι, δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε σαφείς ιδέες, οδικούς χάρτες και προγράμματα συγκεκριμένα. Για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις ε, στην ασφάλεια που όλο και μεταβάλλονται. Για να αντιμετωπίσουμε τις αυστηρές ε, δημοσιονομικές περικοπές των κρατών μελών πρέπει να αντιστρέψουμε την ε, μείωση που συμβαίνει διατηρούμενη των δαπανών και των επενδύσεων. Θα πρέπει λοιπόν οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων να επιβεβαιώσουν και να επαναλάβουν τον Ιούνιο τις δεσμεύσεις των σχετικών Υπουργών Αμήνης δηλαδή 20% των δαπανών για τις ε, δημόσιες αγορές, 35% ε, των δαπανών για εξοπλισμό, 2% για έρευνα και ανάπτυξη και 20% σε συνεργατικά ερευνητικά προγράμματα επιστημονικά. Και θα πρέπει να διατηρήσουμε ε, το... στο επίκεντρο τα αποτελέσματα. Έχουμε το αναθερωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη των αμυντικών ικανοτήτων μας και θα πρέπει βασικός άξονας εκεί να είναι το air surveillance, η εποπτεία του αέρα, η αντιμετώπιση των drones και η πυραυλική άμυνα και και τα θέματα συντήρησης του εξοπλισμού. Διότι αν δεν δούμε ε, πού βρίσκονται τα ελαττώματα, πού βρίσκονται τα προβλήματα και μάλιστα με συνεργατικό τρόπο τώρα, τότε αυτά θα μεταφραστούν, θα γίνουν μεγαλύτερες παγίδες και θα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Όσο λειτουργεί κανείς εθνικά, λειτουργεί κατακαιρματισμένα και αυτό είναι εις βάρος της ευρωπαϊκής άμυνας αλλά και εις βάρος της ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής αμυντικής βάσης πιο συγκεκριμένα το, η στήριξη της βιομηχανίας και η σημασία της έρευνας και ανάπτυξης δεν μπορεί να υπογραμμιστεί αρκετά. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να έχουμε άμυνα χωρίς προγράμματα και δεν μπορούμε να έχουμε προγράμματα χωρίς μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανική αμυντική βάση που να είναι σε θέση και να καινοτομεί και να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, μια συνολική ευρωπαϊκή προσέγγιση χρειάζεται και αυτό περιλαμβάνει θαρρυντικό κανονιστικό ε, περιβάλλον για την άμυνα. Χρειάζεται φορολογικές και χρηματικές πρωτοβουλίες που θα δίνουν κίνητρα, ειδικά για την έρευνα και ανάπτυξη και ε, ανάπτυξη μέτρων που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια κατά την προμήθευση και τον εφοδιασμό. Θα πρέπει να δίνουμε προτεραιότητες και να στηρίζουμε τον ε, κλάδο αυτό, ειδικέ δράσεις. Πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο καθένας θα έχει ίσες ευκαιρίες σε όλη αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πηγή καινοτομίας. Είναι βασικός παράγοντας που διευκολύνει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Βέβαια, χωρίς να πάνε σε έρευνα και ανάπτυξη, οι προσπάθειές μας θα είναι μάταιες αν συνεχίσουν οι μειώσει στι δαπάνε για έρευνα και ανάπτυξη, θα έχουμε λιγότερα αμυντικά συμβόλαια και τελικά οι εταιρείε αυτέ θα μετεγκατασταθούν εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και θα δημιουργούν δουλειέ, καινοτομία, έρευνα, ανάπτυξη αλλού και όχι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και σα δίνω ένα ε, παράδειγμα. Ε, Πυρομαχικά με ε, κατεύθυνση με ασφαλεία, precision guided ammunition θα έρθει αυτή η τεχνολογία σε τρία ή πέντε χρόνια, αλλά σε τρία ή πέντε χρόνια δεν έχουν αξιοποιηθεί αυτοί οι πόροι, θα έχει πάει αλλού. Είναι δεδομένο αυτό, θα έχουν φύγει. Τι πρέπει να, γίνουν. να γίνει λοιπόν, για να ενθαρρύνουμε την έρευνα και ανάπτυξη πρέπει να ενισχύσουμε επενδύσεις σε παραδοσιακή έρευνα προσανατολισμένη προς την άμυνα, σε, με συνεργατικά έργα για έρευνας και ανάπτυξης, με στρατιωτικό σκέλος και πολιτικό σκέλος, με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έρχομαι τώρα για, ε, στις αντιδράσεις για την έρευνα σε σχέση με την κοινή ε, πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Είναι πράγματι πρόκληση αυτό. Και είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ισχυρή πολιτική στήριξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όχι πιο κάτω όμως, οι δράσεις, ε, οι προπαρασκευαστικές δεν θα πρέπει να θεωρούνται υποκατάστατο της εθνικής έρευνας και ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Αμυντική Υπηρεσία έχει σημειώσει σωστή πρόοδο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί. Έχουν καθορίσει τις βασικές παραμέτρους και το περιεχόμενο των δράσεων πρέπει να είναι νέο, προσανατολισμένο προς την άμυνα. Να έχουμε αμυντικές ικανότητες, να έχουμε ατζέντα στρατηγικών ερευνών για να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις και να εστιάσουμε στις πραγματικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής άμυνας. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την διακυβερνητική φύση της αμυντικής συνεργασίας και θα πρέπει να εμπλέξουμε όσο το το περισσότερο τα κράτη-μέλη στην κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη όθεση στα θέματα αυτά ειδικότερα με την πρώτη πρότασή του για τα πιλωτικά προγράμματα για τον τομέα της έρευνας σε θέματα αμήνης. Το πιλωτικό έργο μέχρι το 2016 θα είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική δοκιμή για τους νέους τρόπους με τους οποίους θα εφαρμόζεται η δράση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας και τους νέους τρόπους με τους οποίους θα αξιοποιούνται τα κονδύλια. Θα μιλήσω ειλικρινά. Σε καιρούς λιτότητας είναι εξαιρετικά δύσκολο οι χώρες μέλη να πιστούν να αυξήσουν τις δαπάνες. Παρόλο που η τάση αυτή τίνει να αντιστραφεί σε πολλές χώρες μέλη, πρέπει να ε, προσέξουμε το πόσο ακριβώς θα δαπανίσουμε τα κονδύλια θα πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για να καλυφθούν τα κενά και άρα αν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε συλλογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν δούμε τις ανάγκες μας σε άμυνα, σε, τις αμυντικές μας ανάγκες σε βάθος 15 ετών, καταλαβαίνουμε την ανάγκη ε, συλλογικής ε, δράσης. Ο καλύτερος τρόπος να υπάρχει ευρωπαϊκή αμυντική ολοκλήρωση στην Ευρώπη είναι οι εθνικές ή κατατόπους εταιρείε να συνεργάζονται όλο και περισσότερο μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να δοθούν κίνητρα και εμείς ε, διερευνούμε διάφορα πεδία όπου μπορούν να δοθούν κίνητρα, ακολουθώντας πλήρως την εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ανάπτυξη ε, κινήτρων, για τη συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών πέραν των ε, εθνικών συνόρων των κρατών μελών, τα οποία όμως κίνητρα δεν θα στρεβλώνουν την αγορά. Και θα εξετάσουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Έχουμε το Co-Market, το JD, ε, το, την κατάρτιση για ε, την εξουδετέρωση των ε, αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών π.χ. στην Αυστρία. Έχουμε πάρα πολλά προγράμματα κατάρτισης. Έχουμε και ένα ταμείο θα μπορούσε να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να συγχρονίσουν τον προϋπολογισμό που έχουν για τις επενδύσεις, να λανσάρουν συνεργατικά έργα και προγράμματα, τα οποία από μόνα τους δεν μπορούν να κάνουν το κάθε κράτος μέλος. Το Ταμείο θα μπορούσε αυτό να ε, χρηματοδοτήσει και επιχειρήσει σύμβαση πτώση δράσεις συγκεκριμένες. Και τέλος, σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για ενδεχόμε... μπορεί να υπάρξει στήριξη σε πρόγραμματα διπλής χρήσης τα οποία εμπλέκουν και όλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διπλής εννοείται στρατιωτικής και πολιτικής. Και είναι σημαντικό για δράσεις κοινή πολιτικής ασφαλείας και αμήνης και για την εύρυθμη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Με βάση την εντολή του 2013, εμείς στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Υπηρεσία με πλήρη διαφάνεια συνεργαστήκαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταρτήσουμε προτάσεις που θα παρουσιαστούν στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου με στοχευμένες δράσεις σε ε, π.χ. περιβαλλοντικά πεδία, ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνη στα κράτη-μέλη, διασφάλιση της πρόσβασης στην τεχνολογία και στις βιομηχανικές δυνατότητες, όπως είναι η η βοήθεια σε ορισμένα κράτη-μέλη στα βραχυπρόθεσμα ε, προβλήματά τους και θέματα εφοδιασμού και το καθεξής και ενίσχυση ε, των ευρωπαϊκών συνεργατικών προγραμμάτων. Κάποια παραδείγματα δράσεων που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Αμαντική Υπηρεσία είναι αυτά. Ο δικός χάρτης να λάβει υπόψη του την συμφωνία πλαίσιο της ε, Ευρωπαϊκής Αμυντικής Υπηρεσίας για την ασφάλεια της προμήθευσης του εφοδιασμού μεταξύ άλλων. Από την άλλη πλευρά, σε κανονιστικό επίπεδο τα κράτη-μέλη τόνισαν ότι δεν θα πρέπει να θετηθεί κάποιος νέος κανονισμός και ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε ε, σωστό και συνεκτικό τρόπο εφαρμογής των δύο ε, οδηγιών, την οδηγία για τις δημόσιες αγορές ή κρατικές προμήθειες και την οδηγία για τις ενδοκινοτικές ε, μεταφορές συναλλαγές. Και, <coughs> συγγνώμη, εν ώψη της Συνόδου του Ιουνίου λειτουργούμε συμπερασματικά τα συμπεράσματα του ε, λειτουργούμε συμπληρωματικά, με συγχωρείτε. Τα συμπεράσματα του ε, Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013 είναι αυτό το οποίο καθοδήγησε τη δράση μας. Και τέλος, έρχομαι τώρα στο τρίτο άξονα της ομιλίας μου, που είναι η ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων. Προχωρούμε καλά με το MRDT, ο ενέριος ανεφοδιασμός. Έχει γίνει σημαντική πρόοδος για την δημιουργία μιας ευ... ευρωπαϊκής δομής τάνκερ με πρωτοβουλία των κάτω χωρών και θα μπορεί να αυτό να υλοποιηθεί. Άλλα κρατημέλη βέβαια ενθαρρύνονται να ε, συμμετάσχουν σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Εντοπίζουμε συνέργειες με άλλες χώρες, με το Ηνωμένο Βασίλειο, με τη Γαλλία και εν δυνάμει και άλλους συμμετέχοντες. Έχουμε προτείνει στα κράτη-μέλη που δεν έχουν το Α400 να το αποκτήσουν για να μπορέσουν να κάνουν ένα αέριο ένα ανεφοδιασμό και να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα. Ε, οι χειριστές των Α400 μη μπορούν να αγοράσουν αυτά τα kit για τις πλατφόρμες τους για να ε, πληρούν με τις προϋποθέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Τα συστήματα RPAS μεσαίου υψομέτρου ε, υπάρχουν τηλεκατευθυνόμενα. Και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δουλέψουν περισσότερο σε αυτό το τομέα της πιστοποίησης, της εναρμόνισης ε, των πληρωμάτων και να αξιολογήσουν την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας. Οι μελέτες σκοπιμότητας θα ξεκινήσουν το 2015 και η Ευρωπαϊκή Αμυντική Υπηρεσία μπορεί να διευκολύνει την διάδραση και αλληλεπίδραση με άλλους ενδυνάμει εταίρους για να είναι βιώσιμες αυτές οι επιχειρήσεις, αυτά τα, αυτές οι δράσεις. Όσον αφορά την ολοκλήρωση της κυκλοφορίας, η εργασία για τα μακρόθεν τηλεκατευθυνόμενα αυτά αεροσκάφη βασίζεται στις δράσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας και για τη ΣΑΤΚΟΒ, η επόμενη γενεά των τηλεπικοινωνιών, δορυφορικών τηλεπικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών βρίσκεται υπό την ηγεσία της Ισπανίας ευθυγραμμισμένη με τα σχέδια να υπάρξουν πρότυπα ώστε να προταθούν στα κράτη-μέλη διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Η EDA θα υποβάλει μια τέτοια ε, μελέτη βιωσιμότητας ε, για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ε, με αποτελέσματα που θα είναι διαθέσιμα κατά τέλη του 2016. Κυβερνοεπιχειρήσεις όσον αφορά και την ε, κρυπτογράφηση και κύριες τέτοιες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας ε, βρίσκονται υπό εξέλιξη για την κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και ε, την εξοικείωση με την τεχνολογία. Πρόκειται να δημιουργηθεί μια ένωση για την κυβερνοάμυνα όσον αφορά την αντιμετώπιση hackers. Βρίσκονται υπό εξέλιξη τα σχέδια. Στόχος είναι να προαχθεί η ανάπτυξη της, του δυναμικού άμυνας των κρατών μελών κατά των κυβερνοεπιθέσεων. Ωστόσο από την άλλη πλευρά θα είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένα ενιαίο πλαίσιο συνεργασίας σε σχέση με τα κράτη. Η ευαίσθητη, ο ευαίσθητος χαρακτήρας των κυβερνοεπιχειρήσεων δεν πρέπει να αποτελεί πρόσκομα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, δύο λόγια για την ε, υποστήριξη και τις δράσεις στις υποστηρικτικές. Υπάρχει μία μονάδα υποστηρικτικών δράσεων στην EDA ώστε συστηματικά να παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες όσον αφορά τα σχέδια που αναπτύσσονται μέσα στο πλαίσιο της EDA και τεχνογνωσία. Αυτό σε σχέση με την δράση στην RCA Επίσης ε, στη Λάρισα σε σχέση με το επιτελείο, το, ε, το κέντρο μας στη Λάρισα, RCA ή e TDA από με τα μέσα της ε, κυβερνοάμυνας και έτσι θα πρέπει να υπάρχουν σεμινάρια που θα διεξάγονται και εργαστήρια, καθώς επίσης και στο κέντρο της Λάρισας. Η Λάρισα έχει καλωσορίσει την εγκατάσταση και δοκιμασία και δοκιμές του, λογισμικού σε σχέση με τις, ε, τη δρομολογημένη αυτή δράση καθώς επίσης ε, και θα χρησιμοποιηθούν αυτά μέσα στο πλαίσιο το, της ε, αποστολής στο Μαλί ύστερότερα κατά το 2015. Επίσης μπορεί να παρασχεθεί συνδρομή μέσα στο πλαίσιο επιχειρησιακών δράσεων ώστε να μπορέσουμε να συνδράμουμε όπως έγινε σε σχέση με το 2014. Τώρα στοχεύουμε στο να επικεντρωθούμε στο να μπορέσουν να υποβληθούν προτάσεις για την αγορά εξοπλισμού για υπηρεσίες συγκεκριμένων δράσεων όσον αφορά το πλαίσιο Αθηνά για παράδειγμα. Αυτό ολοκληρώνει την παρέμβασή μου και είμαι έτοιμος να απαντήσω ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Thank you very much indeed, Ms. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντομέκ. Και τώρα ανοίγει η συζήτηση. Ο κύριος Γκάλερ πρώτος παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ντομέκ για την παρουσίασή σας και θα έλεγα, θα έλπιζα ότι το δικό σας επίπεδο φιλοδοξίας μακάρι να ήταν ίδιο με εκείνο το επίπεδο φιλοδοξίας των κρατών μελών μας και των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Η EDA εξυπηρετεί και βρίσκεται στην υπηρεσία των κρατών μελών και των αναγκών τους και εσείς είσαστε ο διαμεσολαβητής για να επιτευχθούν οι προσδοκίες και οι φιλοδοξίες των κρατών μελών. Εσείς θα πρέπει να δώσετε το πλαίσιο για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν όπως πρέπει τα κράτη-μέλη. Πολιτικά πλήρως συμμερίζομαι τη δική σας ε, προσέγγιση ότι η επικείμενη διάσκεψη κορυφής θα πρέπει να ε, αφιερώσει μεγαλύτερο χρόνο στα θέματα άμυνας και όχι μόνο να γίνει μια ε, καταγραφή δυναμικού και υλικού διότι σε σχέση με τα όσα έγιναν το 2013 η παγκόσμια σκηνή, το σκηνικό έχει αλλάξει άρδιν και έτσι δεν μπορούμε απλά να παραμείνουμε σε παροχημένα πλαίσια και επίπεδα και να επαναλαμβάνουμε αυτά τα οποία είχαμε επαναλάβει κατά το παρελθόν και να καταγράφουμε αυτά τα οποία αποφάσισαν οι Υπουργοί Άμυνας κατά τον ε, Μάιο. Θα ζητούσα λοιπόν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να είναι πιο φιλόδοξοι, να έχουν φιλόδοξους στόχους και να χρησιμοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Και να υπάρχει δυνατότητα να κατανοήσουν και να δεχθούν το γεγονός ότι μόνο από κοινού θα είμαστε σε θέση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Μόνο από κοινού μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και να αντέξουμε ως κάτι το εφικτό και δυνατό αυτά που πρέπει δηλαδή ως καθήκοντα να επιτελέσουμε και έργο που πρέπει να επιτελεστεί όπως ταυτοποιήθηκε κατά το πρόσφατο παρελθόν. Διαρωτώ με τώρα και αυτό είναι φυσικά κάτι το οποίο εμείς θα έπρεπε να δώσουμε συνέχεια σε αυτό και να το εξετάσουμε και με τους εθνικούς βουλευτές, ώστε να ασκηθεί πίεση και από πλευράς τους, ώστε να πιεστούν οι κυβερνήσεις να κινητοποιηθούν και να δράσουν. Διαρωτώ με λοιπόν, τι θα έπρεπε να κάνουμε, πού να ασκήσουμε την πίεσή μας αυτή, ένα συγκεκριμένο εξειδικευμένο σημείο σε σχέση με την προκατακτική δράση αναφέρατε για την χρήση δηλαδή έρευνας και τεχνολογίας R&T, Research and Technology, για νέο περιεχόμενο, νέα ε, νέους στόχους για την ανάπτυξη δυναμικού και δεν θα πρέπει αυτό να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο για παράδειγμα, για να υπάρχει εκπλήρωση κάποιων ε, έργων από πλευράς εθνικών προϋπολογισμών. Στόχος είναι να φτάσουμε στο 2% από πλευράς προϋπολογισμών για την έρευνα και ανάπτυξη και τεχνολογία. Πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη να μην θεωρούν επιπρόσθετα προγράμματα της Ευρωπαϊκής, ένα επιπρόσθετο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα υποκατάστατο για μικρότερης εμβέλειας φιλοδοξίες στο εθνικό επίπεδο. Εδώ από πλευράς με, με τους εθνικούς βουλευτές θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Πολύ καλό είναι και είναι θετικό το ότι επισκεφθήκατε τα περισσότερα κράτη-μέλη. Καλό θα ήταν αν μπορούσατε να μας ονοματίσετε και να μας πείτε ποιες χώρες είναι εκείνες που δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα, ώστε να επικεντρωθούμε σε αυτές. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα είσαστε έτοιμος να τις ονοματίσετε και να αποκαλύψετε ποιες είναι. Πιστεύω ότι θα ήταν αναγκαίο λοιπόν να περάσουμε το μήνυμα το οποίο εσείς μας διαβιβάσατε και το μήνυμα το οποίο από τις σταθερές μόνιμες εκθέσεις μας απορρέει και διατυπώνεται ότι πρέπει δηλαδή να δραστηριοποιηθούμε από πλευράς για παράδειγμα Κούκαν και Τάραν σε τις εκθέσεις αυτές που είναι οι πιο πρόσφατες ε, για την χρηματοδότηση αυτών των ζητημάτων που πρέπει να τύχει συνέχεια και να διασφαλιστεί. Ως προς όλα αυτά σας συγχαίρω λοιπόν προπαρασκευάζοντας ε, <clears throat> τη συνάντηση Υπουργών Άμυνας ε, και το, το έργο του Συμβουλίου, κάνατε τη δουλειά σας, ταυτοποιήσατε, εντοπίσατε τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τώρα είναι η δική μας δουλειά να ασκήσουμε πίεση ώστε να προχωρήσουμε περαιτέρω και να επιτευχθούν αποτελέσματα στο Συμβούλιο, <clears throat> ώστε πραγματικά είναι δική μας δουλειά σε σχέση με τα όσα έχουμε εντοπίσει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κούζο παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για το πρόγραμμα αέριο ανεφοδιασμού αναφέρεται την ημερομηνία 2015. Αλλά για να ενεργοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα υπάρχει η καταληκτική ημερομηνία και ακολουθείται ε, το ίδιο σύστημα με αυτό που ακολουθήθηκε με το Α400M. Ως προς την κυβερνοάμυνα και επεκταθήκατε περισσότερο ε, γι' αυτό. Υπάρχουν κυβερνήσεις που ήδη αποκτούν μηχανήματα προσωμείωσης εμπόλεμης κατάστασης, όπως είναι η Βραζιλία για παράδειγμα. Και μετά, τα μη επανδρομένα οχήματα. Είναι κάτι που υπάρχει στο Ισραήλ, από ό,τι είπα, και η Ευρωπαϊκή Άμυνα συνεργάζεται με το Ισραήλ για τα θέματα αυτά. Πώς διαμορφώνεται αυτή η συνεργασία, θα υπάρξει μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας ή θα μας, απλά θα μας κατευθύνουν. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω και εγώ τώρα μια ερώτηση. Σήμερα το πρωί είχαμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες ε, ακροάσεις. Η πρώτη ήταν μια δημοσία ε, ακροάση για τα προγράμματα έρευνας στον τομέα της ασφάλειας. Και ορισμένοι ευρωβουλευτές ε, αναφέρθηκα στις περικοπές ε, στους προϋπολογισμούς έρευνας που οφείλονται και, στο ορίζοντα, και στον ορίζοντα 2020 που οφείλονται ενδεχομένως στην ε, εισαγωγή του σχεδίου Juncker. τι έχετε να σχολιάσετε, ε, δεν βλέπετε κάποιες δυσκολίες Κατά την ενημέρωση μάθαμε ότι το πρόγραμμα αυτό ήταν πρωτοβουλία ουσιαστικά ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. και οι περικοπές ε, στην έρευνα αφορούν και την ασφάλεια αφορούν την ε, έρευνα στον τομέα της ασφάλειας οι οποίες ήταν αρκετά υψηλές μπορείτε να το σχολιάσετε Δεύτερον, είχαμε και ένα εργαστήριο για το pooling and sharing, την ε, συνένωση και την κοινή χρήση. Η γενική ιδέα είναι ότι έχουμε πολλά υποσχόμενα έργα, προγράμματα, αλλά σίγουρα δεν παρατηρούνται και οι καλύτερες δυνατές εξελίξεις. Ε, χρειάζεται να προωθήσουμε και άλλα ε, έργα σε αυτό το τομέα. Είναι δυνατόν να σχολιάσετε. And the third thing our meeting. Και τρίτον, κατά τη συνάντησή μας πριν από αρκετές εβδομάδες αναφέραμε τις, εν λόγω, τις ε, λεγόμενες ε, διοικητικές συμφωνίες μεταξύ της CDA και συγκεκριμένων κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μας αναλύσετε λίγο το ζήτημα αυτό. Να σας ρωτήσω επίσης ε, την κατάσταση συνεργασίας με την Τουρκία στο πλαίσιο της CDA. Να ζητήσω από τον κύριο Ντόμακ να απαντήσει και μετά μπορούμε να επανέλθουμε σε ερωτήσεις και απαντήσεις. Ευχαριστώ. Thank you, Madam ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ επίσης για τα σχόλια και για τις ερωτήσεις. Κύριε Γκάλερ, πρώτα σε εσά. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια που κάνατε σε σχέση με το έργο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας προπαρασκευάζοντας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και γενικότερα τα θέματα της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Αν μου επιτρέψετε να επανέλθω στο συγκεκριμένο ζήτημα της ε, έρευνας και τεχνολογίας και το θέμα των προκατακτικών δράσεων που αναφέρατε. Προβληματίζομαι όταν βλέπω ότι αφενός με την μείωση σε σχέση με τους προϋπολογισμούς για την άμυνα η συνεργασία δεν ήταν ο κανόνας δυστυχώς. Το αντίθετο, το αντίθετο κιόλας. Μειώθηκε, συρρυκνώθηκε η συνεργασία. Η έρευνα και η τεχνολογία και προγράμματα συνέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μόνο στο επίπεδο του 8%. Κατά 7 ποσοστιές μονάδες μειώθηκαν αυτά τα προγράμματα κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ετών. Αυτό είναι πολύ ανησυχητική εξέλιξη στις επισκέψεις μου σε χώρες και αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο επέμεινα και ενέμεινα ιδιαίτερα και το είπα στις αρχικές μου παρατηρήσεις δεδομένου του μεγέθους της υπηρεσίας και των κονδυλίων μας, του δυναμικού μας και πόσο έχουμε προσεγγίσει το έργο μας. Η υπηρεσία πρέπει να αντιμετωπίσει κυρίως τα βιομηχανικά επιχειρησιακά θέματα που αφορούν την άμυνα στην έρευνα και τεχνολογία. Έρευνα και τεχνολογία πρέπει να είναι το επίκεντρο των προβληματισμών και τη δράση μα. και πρέπει αυτή να είναι η πορεία προ μια ισχυρή ενδυναμωμένη ευρωπαϊκή άμυνα. Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, όχι μόνο α, όσον αφορά τι εξαγωγέ μα, αλλά και εσωτερικά και να μπορούμε να είμαστε προπομπή και πρωτοπόροι για να έχουμε ισχυρό πλαίσιο άμυνα, να είμαστε πάροχοι ασφάλεια. Ε, περί αυτού πρόκειται στο ζήτημα αυτό. Να είναι η Ευρώπη αποτελεσματική. Στις επισκέψεις επισκέψεις μου σε χώρες, δεν θα ονοματίσω τις χώρες αυτές, δεν θα αναφέρω ονόματα. Η κύρια αποστολή μου είναι να συλλέξω απόψεις και να συνομιλήσω ειλικρινά και ανοιχτά με τους εκπροσώπους των χωρών που εμπλέκονται εδώ. Αλλά κάποια θέματα με ανησυχούν. Παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες χώρες όπου βλέπουμε ότι τέτοιου είδους δράσεις αντιμετωπίζονται στο συσχετισμό με τις βιομηχανίες άμυνας, για παράδειγμα, για κάποιους λόγους θεωρούνται κάτι που είναι από πλευράς των Υπουργείων Άμυνας ότι είναι θέματα αντιμετώπισης ε, ε, προβλημάτων τριβών, σειράξεων, χωρίς να αντιμετωπίζουν τα θέματα της ανταγωνιστικότητας που πρέπει να διασφαλίζεται για τις ε, βιομηχανίες άμυνας. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να τύχει συνέχεια, όχι μόνο στο επίπεδο βιομηχανιών, αλλά και στα ίδια τα κράτη-μέλη από πλευράς προϋπολογισμών για την άμυνα και Υπουργείων Άμυνας. Εδώ λοιπόν υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν κάποιες χώρες που είχαν κάποια πολιτική στο παρελθόν και τώρα την ανατρέπουν και ξεκινάνε να εξετάζοντας πρώτο λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικές οι βιομηχανίες άμυνας, αλλά είναι πιο σημαντικό για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα θέματα της έρευνας και ε, τεχνολογίας που πρέπει να συνοδεύουν τα ζητήματα άμυνας και να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Ένα άλλο θέμα το οποίο στην ανάπτυξη αυτή θέλω να υπογραμμίσω είναι η αύξηση των κονδυλίων προϋπολογισμών άμυνας που πρέπει να επιτύχουμε. Και εδώ πάλι υπάρχουν προσπάθειες ε, που γίνονται από χώρες σε ένα νέο πλαίσιο άμυνας που πρέπει να μεταφράζονται όμως σε δράσεις υπέρ της ε, έρευνας και της τεχνολογίας. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμα, δεν συμβαίνει. Και επειδή υπάρχουν ελλείψεις ε, πρέπει να επιτευχθούν κάποια πράγματα. Δεν είναι δυνατόν όμως να αναμείνουμε και να καθυστερήσουμε και να περιμένουμε άλλα θέματα να ρυθμιστούν και μετά να σημειωθεί πρόοδος. Άλλες φορές υπάρχει μια πιο εύκολη αναζήτηση λύσης μια δυνατότητα με παραγωγή υλικού αλλού, με αδειοδότηση αλλού, που είναι μια διάμεση λύση, όμως η λύση για την έρευνα και τεχνολογία δεν είναι ο κανόνας, δεν ακολουθείται αυτή η πολιτική ως κανόνας. Και εδώ έχουμε ζητήματα και κονδυλίων που δεν διατίθενται και λόγω της κατάστασης ασφάλειας που επήγει δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Τι πρέπει να γίνει, προκαταρκτικές δράσεις. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε και να εμένουμε για τους δύο μηχανισμούς που λειτουργούν και στα σεμινάρια, τα εργαστήρια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Άμυνας και την ομάδα ε, αξιωματούχων και πραγματογνωμόνων. Ειδική προσοχή, ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται ε, στην αξία που θα έχει αυτό το μέσο ως εργαλείο ώστε να αλλάξει η τροπή των πραγμάτων να γίνει αυτό εκείνο το οποίο θα δημιουργήσει την καμπή προς μια νέα πορεία όσον αφορά την άμυνα και αυτό δεν πρέπει να είναι ποτέ πρόσχημα για μειώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς για την άμυνα αυτό ήταν μέγα σφάλμα πρέπει να επικεντρώσουμε τα προγράμματα σε αυτή την προκατακτική δράση σε ευρωπαϊκή πρόσθετη αξία σε τέτοια προγράμματα και σχέδια πράγματα που θα έχουν νόημα και θα έχουν αποτελεσματικότητα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό είναι εκείνο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και απαντώντας προς την ερώτηση του προλαλήσαντα σε, σχέση με τα τρία ζητήματα όσον αφορά την, τον ανεφοδιασμό ε, αεροσκαφών εν θα ε, πρέπει να γνωρίζετε ότι υπό την ε, ε, ηγεσία της Ολλανδίας ελπίζουμε ότι αυτό το δυναμικό θα μπορέσει να είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά το 2020. Αυτό θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την άλλη μεριά αν, από το αν θα κινηθούμε σε σχέση με τα τρία ή τέσσερα αεροπλάνα που έχουμε υπόψη να χρησιμοποιηθούν τότε όπως το βλέπουμε σήμερα ή αν θα συμμετάσχουν περισσότερα κράτη και ίσως αυξηθεί ο αριθμός των αεροπλάνων εφόσον θα αυξηθούν και οι ανάγκες. Και τότε λοιπόν ίσως θα έπρεπε να προσαρμόσουμε την ε, ε, δράση μας σε αυτό το πλαίσιο. 2020 όμως είναι η ημερομηνία εκείνη κατά την οποία θα μπορούμε να έχουμε αυτή την επέκταση δυναμικού. Για την κυβερνοάμυνα, όπως είπαμε, ε, κάναμε ό,τι μπορέσαμε περισσότερο για την συνειδητοποίηση, την αύξηση της συνειδητοποίησης αυτού του προβλήματος. Περισσότερα πρέπει να γίνουν η περιπλοκότητα είναι ότι δεν είναι πάντα η αρμοδιότητα Υπουργών Άμυνας τέτοια θέματα κυβέρνου άμυνας. Υπάρχει εδώ και η πάρα πολύ ευαίσθητη πτυχή ε, ε, των δεδομένων και της, ε, του δυναμικού. Πρέπει όμως να έχουμε τις δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Ιδιαίτερα με τα ζητήματα τα οποία βλέπουμε ε, υβριδικού πολέμου και κυβερνοπολέμου. Μια πραγματική πρόκληση για το πώς θα πρέπει να διεξάγονται τέτοιες επιχειρήσεις μελλοντικά. Αν θέλουμε να έχουμε επιτυχείς τέτοιες στρατηγικές για τέτοιου είδους πολεμικές αντιπαραθέσεις πρέπει να έχουμε δυνατότητες Υπότιτλοι AUTHORWAVE το πρόγραμμα αυτό να μην αφήσουμε να, να δημιουργήσει κάποιο κενό ή χάσμα σε σχέση με τα κράτη-μέλη μας και να είμαστε πλήρως ανεπτυγμένοι. Σε σχέση με το Ισραήλ, σε σχέση με την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, δεν έχω υπόψη τα σχετικά. Υπάρχουν όμως αρκετοί άξονες ε, εργασίας ε, επί των οποίων ε, αναπτύσσουμε το έργο μας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά βέβαια ότι το Ισραήλ είναι μία από τις χώρες προπομπούς σε σχέση με τις τεχνολογίες όσον αφορά τις ε, τεχνολογίες κυβερνοάμυνας ε, ε, και λογισμικού. Όμως δεν έχουμε εξειδικευμένη τέτοια συνεργασία αυτή τη στιγμή είτε σε τεχνολογική βάση είτε σε λειτουργική βάση με, το, με επιχειρησιακά προγράμματα με το Ισραήλ. Σε σχέση με το άλλο ζήτημα το οποίο θέσατε και το οποίο αναφερόταν στις δυσχέρειες όσον αφορά τα προγράμματα έρευνας για την ασφάλεια και τα όσα παρουσιάστηκαν. Πράγματι, αν δούμε το τι συμβαίνει σε τέτοιου είδους προγράμματα και σχέδια, μπορώ να πω αυτό το οποίο απάντησα στον κύριο Γκάλερ για να σας διασφαλίσω ότι απόλυτα συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες ε, ευρωβουλευτών ε, ως προς ε, τα όσα διατυπώσατε για τις κοινέ το υλικό το οποίο θα συναθρίζουμε και θα επιμερίζουμε pooling and sharing νομίζω ότι πολλά μπορούν να γίνουν. Κάποια πράγματα έγιναν ήδη, δεν έχουν γίνει όμως όλα. Κάποια είναι λιγότερο ευδιάκριτα για το γενικό κοινό σε σχέση με τις δράσεις μας, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα την υπηρεσία άμυνας ως ένα μέσο, ως ένα ε, διαμεσολαβητή αγοράς οπλισμού και εξοπλισμού που αγοράζεται ε, από την υπηρεσία για λογαριασμό κρατών μελών ώστε να υπάρξει κάποια εξοικονόμηση. Όμως το κύριο πρότυπο ή παράδειγμα για το pooling and sharing είναι ο ανεφοδιασμός με καύσιμα εν πτήση. Δείχνονται, καταδεικνύονται εδώ δυνατότητες χρήσης που είναι εποφελείς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, στο σχεδιασμό του προγράμματος, <clears throat> πρώτον, καθορίζοντας τις απαιτήσεις ΟΚΑ τώρα θα λάβει υπόψη και την πλευρά των ε, αγορών μετά από υποβολή προσφορών και η υπηρεσία αγορών ε, θα είναι εκείνη η οποία θα επομιστεί με την, ε, με, την εξέβρεση του πιο εύθετου αυτού ε, υλικού, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και είναι ένα πρότυπο το οποίο μπορεί να τύχει συνέχεια. Θα ήθελα ιδιαίτερα να υπογραμμίσω εδώ κάτι, να τονίσω ότι στο pooling και sharing δεν θα πρέπει να αναμείνουμε να υπάρξουν κάποια προγράμματα από πλευράς όλων των 27 ή όλων των 28 κρατών μελών. Αλλά να υπενθυμίσουμε στα μέλη ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία άμυνας, υπάρχει δυναμικό και μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κρατών μας όπως εκφράζονται και διατυπώνονται. Χρήστες δηλαδή για περιφερειακές ε, τέτοιες δράσεις που θα αποβαίνουν προς όφελος του συνόλου της Ευρωπαϊκής Άμυνας από πλευράς δομών είναι κάτι το πραγματικά θέλω, που πραγματικά θέλω να ενθαρρύνω. Να δίνω κατηγοριοποιημένες ομάδες ε, χωρών, για παράδειγμα στην ε, ομάδα Βάιμαρ από πλευράς Κεντρικής Ευρώπης, από πλευράς χωρών που θέλουν να συνεργαστούν σε αυτές τις συνέργειες, είναι ανοιχτή αυτή η δυνατότητα. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη ως χρήστες και μπορούν να ζητήσουν ε, από την υπηρεσία μας να σχεδιαστούν τα αναγκαία προγράμματα. Το πλαίσιο αυτό λοιπόν από πλευράς υπηρεσίας άμυνας, EDA, πρέπει να ε, μπορέσει να τύχει ευκαιρία ε, τις οποίες θα δραχθούν τα κράτη για να την χρησιμοποιήσουν ώστε να μπορέσουν να ταυτοποιηθούν οι καλύτερες λύσεις, ε, οι βέλτιστες λύσεις και να συναθρήσουμε το δυναμικό όσον αφορά τις δυνατότητες που θα υπάρξουν για να προσφερθούν αυτές οι λύσεις. Τώρα, σε σχέση με τις συμφωνίες, τρεις έχουμε αυτή τη στιγμή όπως θα γνωρίζετε με την Νορβηγία, μία πολύ σημαντικό εταίρος μια συμφωνία πραγματικά πολύ ζωτική ε, ζωτικής σημασίας και όσον αφορά και το πρόγραμμα ανεφοδιασμού εν πτήση των αεροσκαφών έχουμε μια άλλη συνεργασία με την Ελβετία και η πιο πρόσφατη είναι με τη Σερβία που υπεγράφει από την Λέδη Άστον πέρυσι. Τώρα, να αναφέρω κάτι άλλο. Οι διοικητικές αυτές συμφωνίες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υφίστανται Υπάρχουν λοιπόν ως ένα μέσο, ως ένα εργαλείο για χώρες, για χώρες που πραγματικά επιθυμούν να αναπτύξουν το δυναμικό τους που μπορεί έτσι να γίνει λειτουργικό, διαλειτουργικό και να συνδυάζεται με το δυναμικό των ευρωπαϊκών χωρών. Και ταυτόχρονα να υπάρχει ανάπτυξη κοινού δυναμικού. Να μην έχουμε υπόψη να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς αυτά τα δυναμικά, αυτές οι συμφωνίες διαπραγματευόμαστε και σήμερα είχα πραγματικά την αρχική πρώτη συνάντηση με τις Ουκρανικές αρχές. Είμαστε σε διαπραγμάτευση με τους Ουκρανούς για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις αυτές, για να προχωρήσουμε με μια το δυνατόν νωρίτερη ε, προώθηση αυτής της συμφωνίας που θα εξεταστεί υστερότερα, μεταγενέστερα εφέτος. Εν πάση περιπτώσει και πάλι εδώ μπορούμε να δούμε το τι θα ενταχθεί στην διοικητική συμφωνία, που είναι σε μεγάλο βαθμό κάτι το οποίο τα κράτη-μέλη πρέπει τα ίδια να εγκρίνουν, αλλά και από την άλλη πλευρά φυσικά με ομοφωνία να εγκρίνουν, αλλά και για τομείς ενδιαφέροντος που θα ενδιαφέρουν και θα είναι ενδιαφέροντες αμφωτέρωθεν και για την χώρα που θα θέλει να συνάψει μια τέτοια συμφωνία μαζί μας αλλά και για τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Αυτά σε σχέση με την κατάσταση για αυτό το θέμα, για τις σχέσεις μας με την Τουρκία όπως πολύ καλά γνωρίζετε η διοικητική συμφωνία που βρίσκεται υπό εξέταση έχει παγώσει, έχει τροχοπεδηθεί αυτή τη στιγμή και δεν, δεν προχωρεί. Αν υπάρξουν θετικές εξελίξεις που θα μας επέτρεπαν να δώσουμε συνέχεια και να κινηθούμε προς την επίλυση των ε, ε, εκκρεμούντων προβλημάτων, τότε εντάξει θα είχαμε τη βούληση να προχωρήσουμε. Αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή και έτσι έχουν παγώσει τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ζητήσω να διευκρινίσετε κάτι που αφορά την πρωτοβουλία της Κεντρικής Ευρώπης. Είναι πολιτικός οργανισμός. Είναι μια ομάδα ομάδα αυτή η πρωτοβουλία. Μπορείτε να μας αναλύσετε λίγο το θέμα αυτό της συνεργασίας στο πλαίσιο αυτής της πλατφόρμας, διότι κάποια κράτη που είναι μέλη της δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ε, όπως είπα, η συνεργασία είναι με κράτη που έχουν συμφωνίες Και αυτό είναι που θα ζητηθεί σε αυτές τις ομάδες. Υπάρχουν πρωτοβουλίες που ορισμένε φορές ε, όσον αφορά τις δυνατότητες δεν συμπεριλαμβάνουν όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις. Uh, would you like... Εκτός μικροφώνου, κυρία Πρόεδρε. Όπως φαίνεται τα μέλη εδώ της αίθουσας είναι ικανοποιημένα με τις απαντήσεις. Αλλά έχετε το ελεύθερο να κάνετε παρατηρήσεις ε, αν θέλετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Παραμένω στη διάθεσή σας και μπορώ να επανέλθω μετά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. το οποίο ελπίζω να ικανοποιήσει τις φιλοδοξίες που χρειάζεται η άμυνα στην Ευρώπη σε τόσο δύσκολες εποχές με όλα τα γεγονότα, σε όλα τα σημεία του κόσμου και σε ένα σωρό χώρες. Είμαι στη διάθεσή σας λοιπόν για να επιστρέψω εδώ για να ξανασυζητήσουμε όποτε το επιθυμείτε. I ε, με ειδοποιήσε η κυρία Γιάννη ήθελε. Όχι, συγγνώμη. Δεν κατάλαβα σωστά. Ε, αξιότιμη κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερος ε, για την παρουσίαση αυτή. Είναι βέβαιο ότι θα παραμένουμε σε έπαφη και με μεγάλη μας χαρά θα σας ξαναπροσκαλέσουμε σε συναντήσεις μετά από το Συμβούλιο, το επόμενο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Να σε ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 28 Μαΐου συνάντηση δηλαδή της ε, Υποεπιτροπής ΣΕΔ. Η σημερινή συνάντηση με αυτή την ανακοίνωση τερματίζεται. Ευχαριστώ πολύ.